Well, welcome everybody and thank you for being here. Καλώς ήρθατε όλοι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος αυτό το εργαστήριο για την ε, μείωση των ε, εκπομπών μη διοξιδιού του άνθρακος. Ξεκίνησε όλη η προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Αρχίσαμε να εξετάζουμε τους υδροφλουράνθρακες. HFC23, 123. Και τι ανακαλύψαμε. Ότι οι εκπομπές εκτός διοξιδίου του άνθρακος δεν αντιπέζονται το ίδιο με τις εκπομπές του του άνθρακος ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό μπορεί να έχει δίνει σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση του κόστους των πολιτικών για το κλίμα και αύξηση του ρυθμού της κλιματικής πολιτικής χωρίς να χρειάζεται μια παγκόσμια συμφωνία, συμφωνία σε παγκόσμια διάσταση. Στη διαστάσεις που είχαμε υπόψη μας στην Κοπενχάγη. Και ξέρουμε τώρα πια ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ξεκινήσαμε το εξετάζουμε το θέμα με συναδέλφους, όπως με τη Λίνα Μακιούαν, τον κύριο Ζέμπερ και άλλους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε, πρέπει να καλύψουμε πολλά για να δημιουργήσουμε πολιτική ευρωπαϊκή και παγκόσμια όσον αφορά τις εκπομπές εκτός διοξιδίου του άνθρακος. Να είμαστε πολύ αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι στις προσπάθειές μας δεν είναι οι αγαπημένες λέξεις στην περιβαλλοντική πολιτική αυτές. Οι λέξεις ευαίσθητη πολιτική, ευαίσθητη πολιτική, περιβαλλοντικά φιλική, βιώσιμη, αυτές οι λέξεις μας αρέσουν. Αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως στην περιβαλλοντική πολιτική. Ε, εγώ θα έλεγα ότι είμαι άνθρωπος σχολείται με τα περιβαλλοντικά με υπολογιστή. Θα ήθελα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διότι το θέμα της αλλαγής του κλίματος είναι τεράστιο και χωρίς αποδοτικότητα δεν μπορούμε να ανηκήσουμε. Χωρίς αποτελεσματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ας ξεκινήσουμε μετά από αυτό και να δώσουμε το λόγο στην Λίντα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, διότι ο συνήθως το κοινοβούλιο ξεκινάμε αργά. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή παρουσίαση από εμπειρογνώμονες, διότι εμείς σαν πολιτικοί καθόμαστε εδώ και ακούμε τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωπικού μας. Το να είναι τόσο, τόσοι πολλοί εξωτερικοί εμπειρογνώμες παρόντες είναι πολύ χρήσιμο. Πάντα εστιαζόμασταν στο δεξί του άνθρακα. Μιλούσαμε για το δεξί του άνθρακα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα αέρια του θερμοκηπίου και όσο μειώνονται τα επίπεδα διοξιδίου του Άνθρακο πρέπει να ρυθμίσουμε και τα ποσοστά των άλλων αερίων για να πετύχουμε τους στόχους περικοπής των εκπομπών. Καλωσορίζω λοιπόν αυτό το εργαστήριο. Έχουμε προφορική ερώτηση και ψήφισμα την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλει να προωθήσει το Κοινοβούλιο και να αναλυθεί η δράση. Και χαιρόμαι που είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει και αυτή την άποψή της και τι μπορούμε να κάνουμε και περιμένω να ακούσω τους εμπειρογνώμονες. Α, συγγνώμη. Έλεγα ότι ξαναπήρατε την Προεδρία. Έχουμε το πρώτο τμήμα, το θέμα των εκπομπών εκτός δεξιού του άνθρακος, Dr. Neil Harris, ο πρώτος ομιλητής μας, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, θα μιλήσει για τη σχέση που άρχισε μεταξύ μειώσεως της θηβάδας του όζοντος και της αλλαγής του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ τους Προέδρους τη συνεδρία αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου με κάλεσαν να έρθω εδώ και να μιλήσω σε αυτή τη συνάντηση. Ξέρω ότι είσαστε πολύ άσχολοι στην Ευρώπη και χαίρομαι που παρόλα αυτά ε, εξετάζετε και μέσω μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπου μια ταχεία δράση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά, μακροπρόθεσμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα μιλήσω για την επιστήμη πίσω από κάποια από τα αέρια εκτός ε, διοξιδίου του άνθρακος και σωματίδια. Ε, καταρχάς, να αναφερθώ στην αλλαγή του κλίματος τα επόμενα χρόνια και την ταχύτητα με την οποία γίνονται διάφορες αλλαγές στο κλίμα. Θα αναφερθώ στα τέσσερα αέρια, θα αναφερθώ στο όλο ιστορικό όσον αφορά τη λογική που ακολουθήθηκε για να εφαρμόσουμε μέτρα που θα κάνουν τη διαφορά βραχυπρόθεσμα και θα ολοκληρώσω με συμπεράσματα και τις διαφορές που θα διαπιστώσουμε. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα, πάνω αριστερά, βλέπετε έξι πιθανότητες όσον αφορά τις αλλαγές του κλίματος. Φαινόμενα που θα μπορούσαν συμβούν πάρα πολύ γρήγορα, ανάλογα με τη θέρμανση. Δυτική, ανταρκτική, ε, παγετώνας της ε, Γρυλανδίας, αρκτική, πάγο θερινό, θα μειωθούν κατά 50% με τα μέτρα αυτά που έχουν συμφωνήσει. Έχουμε δυτική, ε, το λιώσιμο των πάγων της Δυτικής Αρκτικής... και επίσης και τις αλλαγές όσον αφορά την κυκλοφορία των διαφόρων ρευμάτων. Βλέπετε ότι λένε ότι είναι σταδιακή η αλλαγή με την αύξηση της ε, θερμοκρασίας ε, δύο βαθμών με την παρό του χρόνου και ότι οι αλλαγέ κατά κάποιο τρόπο είναι ευχάριστε. Αυτό που θα δούμε πέραν από τη σταδιακή αλλαγή θα είναι ταχεία άφηξη γεγονότων και ακραία γεγονότα, φαινόμενα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε στην αρχή για να μειώσουμε του ρυθμού αυξήσεω τη θερμοκρασία ή τη αλλαγή του κλίματο είναι κάτι πολύτιμο. Γιατί έτσι κερδίζουμε χρόνο για να προετοιμαστούμε για τα συνέπειε των αλλαγών Έγινε πρόσφατα ένα εργαστήριο. Το οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και εξέτασε κάμια από αυτά τα θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη. Βλέπετε ε, το στρώμα πάγου της Γρυλανδίας που λιώνει, την αλλαγή στην κυκλοφορία των διαφόρων ρευμάτων και τους παγετώνες της Άλπης ε, που, θα, που τα τελευταία 100 χρόνια λιώνουν πάρα πολύ γρήγορα είναι παγκόσμια θέματα πάρα πολύ σημαντικά και χρειάζονται και επίσης έχουμε κάποια θέματα που είναι καθαρά ευρωπαϊκά. Αυτό το γράφημα είναι πολύ μικρό για την αίθουσα αυτή για να μπορέσετε να δείτε. Εξηγώ με τα τοξάκια, με τα βελάκια, είναι από την έκθεση τα IPCC. Την τελευταία έκθεση του 2007 τα IPCC και πάνω βλέπετε ε, τι γίνεται με τις εκπομπές του εξιδίου του άνθρακος το 2005 και δεξιά βλέπετε θετικές και αρνητικές τιμές αριστερά. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη συνιστόσα αλλαγή του κλίματος. Μετά βλέπουμε το μεθάνιο που είναι περίπου έχει μισό το αντίκτυπο του διοξιδίου του άνθρακος. Έχει μεγάλη συνέπεια από μόνο του το μεθάνιο και μπορούμε βραχυπρόθεσμα να το αλλάξουμε, αλλάξουμε το στο μεθάνιο. Πιο κάτω έχουμε τα HFC και τα λογόνα άνθρακος. Λοιπόν, θέλουμε να σχεστούμε τα HFC. Τα HFC έχει πολύ μικρή, ε, μικρό αντίκτυπο. Δεν έχει επηρεάσει πολύ την ατμόσφαιρα. Μπορούμε να σταματήσουμε την αύξηση των συγκεντρώσεων του αερίου αυτού. Ε, ούτω ώστε να μεγαλώσει με τα ανθρακούχα. Μετά έχουμε ρηπαντές που οδηγούν στη διαμόρφωση ε, διαφόρων σωματιδίων και κάτω βλέπετε τι γίνεται με το μαύρο άνθρακα που αλλάζει. Δεν βλέπετε τα σωματίδια και τα αεροζόλ που να διαχωρίζονται έτσι. Ψύχουν περισσότερο. Ο μαύρος άνθρακας δημιουργεί τοπικό αντίκτυπο. Θα το πούμε σε λίγο αυτό. Βλέπετε πως το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ ωφέλησε την, το, πρόβλημα της μειώσεως στη βάδα στο ζώντα. Πάνω βλέπετε κίτρινο πορτοκαλί. Βλέπετε πως άλλαξαν οι εκπομπές από το 80 μέχρι το 2020 με προβολή, με μεγάλη μείωση των εκπομπών σε αυτή τη φάση. Το κάτω γράφημα ε, δείχνει τη συγκεντρώση στην ατμόσφαιρα που μειώνονται με πιο αργούς ρυθμούς από τις εκπομπές, διότι μένουν για 100 ε, χρόνια περίπου στην ατμόσφαιρα. Περίπου, ε. Γι' αυτό το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ ήταν κάτι επιθυμητό και δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Βλέπετε το γράφημα. Δεξιά βλέπετε ποια είναι η συνέπεια του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ στην αλλαγή του κλίματος ε, στο πάνω γράφημα, στην πάνω γραφική παράσταση βλέπετε την αντίστοιχη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα που θα προέρχεται από CFCs. Θα μπορούσαμε αν είχαμε υπολογιστάκια να υπολογίσουμε τα διάφορα αέρια και τη συνδρομή τους. Κάνοντα σύγκριση βλέπουμε ότι το κίτρινο μειώθηκε όσον αφορά τον αντίκτυπο στο κλίμα και πολύ απότομα μειώθηκε τα τελευταία 10-15 χρόνια. και δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την ακτινοβολία, επίδραση στην ακτινοβολία και στην αλλαγή του κλίματος. Στο γαλάζιο κομμάτι βλέπετε τι έχουμε εξοικονομήσει από, εν συγκρίση με την συνεχή αύξηση χρήσεως των CFCs, χωρίς μείωση που θα που επιτυχάνεται μέσω του πρωτόκολλου του Μοντρεάλ. Αυτό που δεν βλέπετε πάνω είναι δύο γιγατόνι άνθρακα που είναι ο στόχος ε, του πρωτοκόλλου του Κιώτο για το 2018 αυτή η εξοικονόμηση. Οι εξοικονομήσεις από το CFC ήταν 10 με 12 γιγατόνι άνθρακα. Το πρωτόκολλο του Μόντρεάλ ήταν 5-6 φορές ο στόχος του Τόκιο από το 2008 μέχρι το 2012. Βλέπετε πόσο επιτυχές ήταν και έχει και παράπλευρα αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση θερμοκρασίας στον κόσμο και την αλλαγή του κλίματος. Τα HFCs είναι τα στοιχεία που βλέπετε στο, κάτω γράφημα αριστερά. Ε, βλέπετε το, τη μείωση του όζοντος. Στον κάτω άξονα βλέπετε πόσο με ποιου ρυθμού, πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα στοιχεία στη μείωση του όζοντα. Τα HFC δεν μειώνουν το όζον και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν σαν υποκατάστατα για τα CFCs και τα HCFCs ε, διότι οι εκπομπές τους έτσι περιοριζόταν. Αν κάνεις παρόμοιο υπολογισμό όσον αφορά τι δυνατότητε αλλαγή του κλίματος, αύξηση θερμοκρασία, βλέπετε ότι τα HFCs έχουν μεγάλη δυνατότητα να αύξηση θερμοκρασία. Με, μεγαλύτερο αντίκτυπο. Περισσότερο από τα CFCs που είναι πάνω τα τρία γραφήματα. Οι προβολές που κάναμε τι δείχνουν. Ο, ότι η αύξηση αντιστοιχούσε τον HCFC σε άλλα 9 γιγατόνους άφακο το χρόνο ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Σημαντικές συνιστώσεις λοιπόν αυτά τα στοιχεία στην αλλαγή του κλίματος. Αυξάνεται ε, η, συμμετοχή τους πολύ γρήγορα. Βλέπετε από το Cape Grim στην Τασμανία το γράφημα αυτό και δείχνει πόσο το SFC 1 2 1234α που χρησιμοποιείται στο εγκληματισμό ε, των αυτοκινήτων αυξήθηκε από το 2008. Από 0 πήγαμε στα 45 ε, τμήματα ανά τρισεκατομμύριο. Αν γίνουν περικοπές αρχικά με σημαντικές, θα σταθεροποιούνταν οι συγκεντρώσεις και ο αντιχτύπος στο κλίμα. Αυτό είναι το βασικό με τα HCFC μπορείς να κόψεις, να εκριζώσεις το πρόβλημα πριν φουντώσει. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η πρόκληση για τα HFCs. Λοιπόν, αναφέρθηκα στο, στη Μαύρη Θάλη, έγινε μια έκθεση για το τροποσφαιρικό όζον και το μαύρο άνθρακα, πρόσφατα μια έκθεση, μια δύο από τις διαφάνειές μου φίλους αυτό. Ο μαύρος άνθρακας είναι μαύρος και απορροφά το φως. Άρα θερμαίνει την ατμόσφαιρα. Και όταν πέσει στο πάγο ή στο χιόνι, σκουραίνει το σιόνι και το πάγο, άρα λιώνει πιο εύκολα ο πάγος και το χιόνι. Άρα έχουμε ατμοσφαιρικό αντίκτυπο, το μαύρο άνθρακα όταν είναι στην ατμόσφαιρα, αλλά αν εκπέμπεται κοντά σε λευκές περιοχές, παγετώνες κλπ, έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτές τις ε, περιοχές. Η διάρκεια ζωής του μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι ε, μέρε με εβδομάδε. Δεν κρατάει πολύ στην ατμόσφαιρα. Οποιασδήποτε αλλαγέ λοιπόν στις εκπομπές ε, θα έχουν άμεσα αποτελέσματα σχεδόν. Αντίθεση με, το, με τα HFC, όπου ποια είναι η λογική. Περικοπές τώρα για τι εκπομπέ για να μην επιδεινωθεί το πρόβλημα, εδώ σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε άμεση μείωση α, ε, στις, στις συνέπειες που έχει όσον αφορά την απορρόφηση του φωτός κλπ. Εδώ βλέπετε πώς το ο όζον στο FIU στη Ελβετία αυξήθηκε από το 1985 ε, μέχρι τώρα. Αυξήθηκε, σταθεροποιήθηκε και ενδεχομένως τα τελευταία χρόνια να μειώθηκε κάπως. Οι ρηπαντές, μεθάνες και μεθάνιο και ε, οδηγούν στη μείωση του όζοντα. Δεν έχει συμφωνηθεί, θα μπορούσε να ελεγχθεί αυτό με εμείς των ρηπαντών. Το τροποσφαιρικό όζον διαρκεί περίπου εβδομάδε αυτήν τη διάρκεια ζωή του. Αν μπορούν να γίνουν αλλαγέ εκπομπών και πάλι, άρα η ανταπόκριση είναι αρκετά γρήγορη. Δηλαδή, το όζον σε ένα χρόνο περίπου δεν θα επηρεάζεται πια από τις σημερινές εκπομπές. Μεθάνιο βλέπουμε στο πάνω διάγραμμα πώς συγκεντρωνόταν την τελευταία 30 αυξήθηκε, σταθεροποιήθηκε λίγο τα τελευταία χρόνια και δείχνω τη αλλαγή του όζοντα, αριθμούς ανάπτυξης ε, χρόνο με το χρόνο. Το μεθάνιο, όπως σας έδειξα πριν, είναι ε, πολύ σημαντικό για τα φαινόμενα θερμοκηπίου και δημιουργεί ε, τροποσφαιρικό όζον. Έχει, είναι περίπλοκες οι πήγες, μερικές είναι φυσικές, μερικές ανθρωπογενείς, Γεωργία Φερρυπίν, είναι σημαντική πηγή, από άνθρακα, από πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Το μεθάνιο διαρκεί 10 χρόνια, έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Αν οι εκπομπές μειωθούν, η ανταπόκριση ατμόσφαιρας θα είναι μετά τα μερικά χρόνια. Πολύ κάτω από την κλίμακα του ενός αιώνα που είναι η ανταπόκριση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Εδώ λοιπόν ένα γράφημα από δέξη Γιούνα για το μαύρο άνθρακα και το τροποσφαιρικό όζον. Αριστερά βλέπετε τις ιστορικές υψηλές θερμοκρασίες, μετά από εκεί έχουμε τέσσερις γραμμές που αφορούν το μέλλον. Η πάνω γραμμή είναι η συνήθις υπόθεση. Βασίζεται σε γνωστούς ελέγχους των διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου. Η επόμενη γραμμή πιο κάτω δείχνει τις πιστευτές αλλαγές του διοξείδου θα άνθρακο σας αποκαλώ. Πιστευτές, αποδεκτές, πιθανές. Μέχρι το τέλος του αιώνα, 2050 τουλάχιστον, έχουμε μείωση στη θέρμανση περίπου μισό βαθμό. Αν δείτε τις επόμενες δύο γραμμές, δείχνουν τα αποτελέσματα των μέτρων σε αυτό το μεθάνιο και το μαύρο άνθρακα για την αλλαγή του κλίματος. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι παρόμοια σε τάξη μεγέθους και μπορούν όμως να λάβουν χώρα νωρίτερα. Αν θέλεις λοιπόν να καθυστερήσεις ή να μειώσεις την πιθανότητα ταχαίων αλλαγών του κλίματος και να καθυστερήσεις και την ε, πιο σταδιακή αλλαγή. Αυτά πρέπει να έχει υπόψη σου. Είναι η πρώτη υποψήφη. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Κάποιε συνέπειε τη αλλαγή του κλίματο συμβαίνουν σταδιακά, άλλε αλλαγέ γίνονται πιο γρήγορα. Κάποιε από τι γρήγορε αλλαγέ θα μπορούσαν να είναι αρκετά δραματικέ, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτέ είναι και πιο δύσκολο να προβλεφτούν. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η μετάβαση τις επόμενες δεκαετίες και ποια θα είναι η τελική κατάσταση. Αυτό είχαμε υπόψη μα. Εμεί ε, ε, οι επιστήμονε. Αν έχουμε μια ατμόσφαιρα διπλάσιο του άνθρακο. Το Μόντρεαλ, το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ήταν πολύ επιτυχέ στα μέτρα όσον αφορά τη μείωση των αερίων ε, θερμοκηπίου, θετικά αποτελέσματα αλλαγή του κλίματο και έλεγχο μεθανίου, μαύρου άνθρακα και τροποσφαιρικού όζοντα, που είναι πρόδρομε ουσίε, θα μπορούσαν να κάνουν ε, σταδιακά βραχυπρόθεσμα αλλαγέ για την αλλαγή του κλίματο. Βραχυπρόθεσμα τι εννοώ, 5 με 20 χρόνια και όχι ότι έχουμε υπόψη όταν, λέμε, όταν μιλάμε στο πολιτικό πλαίσιο, όταν λέμε κάτι ότι είναι βραχυπρόθεσμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι να σκεφτόμαστε και κύκλους, έτσι, και υπάρχουν και κοινοβουλευτικοί θητείες και καλό είναι να νομοθετούμε πριν τελειώσει. Ο κύριος Μάρκο Γκονθάλες, Γενικός Γραμματέας του Πρωτοκόλου του Μόντρεαλ, θα μιλήσει ε, για τις ε, συνέργειες των ε, κυβερνήσεων και το πρωτόκολλο του Κιώτο. Πολλές φορές ακούμε να λένε οι συνάδελφοι ότι δεν λειτουργούν οι διεθνείς συμφωνίες, μπορούν να λειτουργήσουν και το πρωτόκολλο του Μόντρελ είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Uh, thank you σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή την παρουσία μου εδώ σήμερα. Θα ήθελα να πω για την ιστορία ότι είχα διατελέσει βουλευτή στο Κοινοβούλιο της Κώστα Ρίκα ε, στις αρχές δεκαετίας του 90. και εκεί μας απασχολούσαν θέματα του όζοντος, η έκπληση του όζοντος, προστασία της τυφάδας του όζοντος, βιοπικιλότητα. Έκτοτε έχουν παρέλθει πάνω από δύο δεκαετίες και είμαι ενώπιόν σας και είναι μεγάλη τιμή αυτή που αισθάνομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλώ με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος συγκεκριμένα και μάλιστα να είμαι στο πάνελ αλλά και ε, να έχουμε και την ευκαιρία να συζητούμε δημόσια. Like to, to Θα ήθελα από την αρχή και εκ των προτέρων να καλωσορίσω αυτή την πρωτοβουλία το μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι αυτή η συνολική σφαιρική προσέγγιση είναι πάρα πολύ απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Έχω διπλή ιδιότητα και θα χρησιμοποιήσω και τις δύο μου ιδιότητες στην παρουσίαση. Θα σας μιλήσω και προσωπικά, θα σας εκθέσω τις προσωπικές μου απόψεις για το θέμα, αλλά επίσης θα μιλήσω ως εκτελεστικός γραμματέας του πρωτοκόλου του Μορεάλ. Ελπίζω να καταλάβετε όλοι σας πότε θα μιλώ προσωπικά και πότε θα μιλώ με την άλλη μου ιδιότητα. Um, uh, και επίσης, όπως είπε ο καθηγητής κύριος Χάρης, νομίζω ότι δεν χωράει καμία αμφιβολία και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ε, ότι αλλάζει το κλίμα. Και ε, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει κλιματολογικά. Ωστόσο, υπάρχουν και οικονομικοί παράγοντες και πολιτικοί που αφορούν την εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν ή των όσων θα συμφωνηθούν στο μέλλον. Αυτό είναι μια πρόκληση πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ περίπλοκη. Αυτό τον καιρό γίνονται διαπραγματεύσεις που μας δείχνουν πως έχει κατάσταση. Συμφωνώ πάρα πολύ με σας τους δύο ε, του Πρόεδρους, στην εισαγωγή σας ότι τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια κλιματική πολιτική ε, αφορούσε τα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν μακρά διάρκεια και το διοξίδιο του άνθρακα. Όπως γνωρίζουμε, ε, άνθρακας υπάρχει παντού στη γη. Ακόμα και στο DNA και τις πρωτεΐνες και στα συστατικά κάθε είδους ζωής. Αν δεν υπήρχε άνθρακας, δεν θα υπήρχε ζωή η ίδια στη γη. Ε, here. Ε, με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε. Οπότε δεν μας εκπλήσει ότι βρίσκουμε τον άνθρακα στην καρδιά του σύγχρονου πολιτισμού μας. Και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σωστά εντοπίστηκαν ως κύριος ένοχος της κλιματικής αλλαγής και συνεργάζονται οι θύνοντε ε, του κόσμου για το πρωτόκολλο του Κιόπτο για να προσπαθήσουν να μειώσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν. Μέχρι πρόσφατα όμως έχει δοθεί πολύ λιγότερη προσοχή σε άλλους ρηπαντέ πλην διοξιδίου του άνθρακα. Ε, μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει κανείς να δίνει περισσότερη σημασία και προσοχή σε αυτό το παράγοντα. Και οι πολιτικές μας. Αυτό δεν μας εκπλήσει καθόλου, διότι σε έναν κόσμο που διέπεται από την οικονομία ο κόσμος περιμένει απόδοση των μέτρων, είτε πρόκειται για εθνικούς είτε για διεθνείς παράγοντες. Και με τον ίδιο γνώμονα οι πολιτικές ακριβώς αυτό αποσκοπούν, με ειδικούς μηχανισμούς, ειδικούς θεσμούς, με διμερείς συμφωνίες, διμερεί προγράμματα ή πολυμερεί, με στόχο ακριβώς αυτόν. Οπότε, μια συνολική ε, πολιτική θα πρέπει να επιταχύνει την παγκόσμια απόκριση στην κλιματική αλλαγή. Αυτή όμως η απόκριση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένα εναλλακτική ε, λύση στα όσα ήδη κάνουμε. Όχι, συμπληρωματική, ακριβώς για να έχουμε συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής, ε, βράχη πρόθεσμα και να την καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά. Για να το πω με δύο λόγια, στόχος των διαφόρων προσπαθειών και των εντολών που έχουμε, που κάνουμε ό,τι μπορούμε και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και μάλιστα το συντομότερο, θα πρέπει να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Οπότε έχει μεγάλη σημασία ακριβώς συνεργασία και συνέργειες. Τι θα πει αυτό. Συνέργεια τι είναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε στην παγκόσμια διακυβέρνηση και είναι ε, στον πυρήνα και στην ουσία ε, των συζητήσεων για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Και θα πρέπει να είναι και ε, μια αρχή που να διέπει τις συζητήσεις μας για την κλιματική αλλαγή και στον ΟΗΕ. Βλέπετε ήδη από την εισαγωγή ότι χρησιμοποιώ και τις δύο μου ιδιότητες. Επιτρέψτε μου τώρα να επικεντρωθώ στη σύμβαση της Βιέννης και στο πρωτόκολλο του Μοντρεάλ σε σχέση πάντα με την κλιματική αλλαγή. Πώς γεννήθηκαν αυτές οι συνθήκες για το περιβάλλον. Ήταν μικρή αλλαγή η αρχή, μάλλον 24 χώρες στην αρχή, στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, με στόχο να μειωθούν ε, οι εκπομπές μόνο ε, στις αναπτυγμένες χώρες και αυτό φορούσε δύο είδη ουσιών. 50% ε, σήμαινε μείωση και όχι 100% στην αρχή της ισχύω. Και σιγά σιγά εντάθηκε η προσέγγιση, ενισχύθηκε και καρποφόρησε μετά από τα δεδομένα που είχαμε, τα επιστημονικά, τα σύγχρονα. Και μάλιστα αυτό δεν το είχαν φανταστεί, δεν το είχαν ονειρευτεί, ούτε κάνει πιο αισιόδοξοι των αρχικών διαπραγματευτών. Αυτή η προσέγγιση του Μοντρεάλ ενισχύθηκε και βασίστηκε σε επιστημονικά στοιχεία και τελικά ήταν και πολύ αποδοτική και πάρα πολύ αποτελεσματική και επιτυχημένη. Μέχρι σήμερα έχουμε συνολική μείωση πάνω από 97% των ιστορικών επιπέδων ε, κατανάλωσης ε, όλων των ε, βλαβερών ουσιών και εκπομπών. Και μαζί με τη Σύμβαση της Βιέννης είναι οι μόνες συμβάσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών που κατάφεραν να ε, επιτύχουν παγκόσμια κύρωση. Και όπως γνωρίζουμε, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα. Και σε όλα τα κράτη του κόσμου σήμερα συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ε, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και αλλαγές. Άλλο σημαντικό τώρα επίτευγμα του πρωτοκόλου του Μόντρεαλ που γνώρισε ευρύτατη ε, αναγνώριση ήταν, όπως είπε και ο καθηγητής Χάρης, η συνεισφορά των μερών της σύμβασης του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για την προστασία του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής. Γιατί δεν είναι μόνο το αέρια του θερμοκηπίου, είναι και άλλες ουσίες που εκπλήουν τη στιβάδα του όζοντος και τελικά Είχαμε τεράστια αποτελέσματα ευεργετικά, όχι μόνο για τη στιβάδα του όζοντος, αλλά και για το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. You to explain. I will also... Όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω προηγουμένως, με τις τρεις αυτές γραφικές παραστάσεις που βλέπετε στην οθόνη, το κέρδος που είχαμε από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, από μείωση ε, των εκπομπών ε, που οδηγούν σε κλιματικές αλλαγές, η αποτροπή, η πρόληψη. Αυτά τα τρία γραφήματα, οι γραφικές παραστάσεις είναι ίδιες, αλλά μετρούν διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο μετρά τη μάζα, το βάρος των εκπομπών και όλο αυτό το γαλάζιο τμήμα είναι τι καταφέραμε να προλάβουμε, να αποτρέψουμε. Το δεύτερο είναι εκπομπές που εκπλήγουν τη στιβάδα του όζοντος. Δηλαδή καταστρέφουν ουσιαστικά. Και βλέπετε ένα γαλάζιο πεδίο αριστερά το οποίο αντιπροσωπεύει τη σωρευτική μείωση ή αποτροπή όλων των ε, βλαβερών εκπομπών αερίων που θα μπορούσαν να έχουν επιδράσει αρνητικά στο κλίμα. Και το τρίτο είναι το πιο ενδιαφέρον ίσως ως γραφική παράσταση. Αν κοιτάξετε το ε, ανοιχτό πράσινο στο πάνω μέρος της ε, γραφικής παράστασης είναι οι ιστορικές ε, λεγόμενες εκπομπές της δεκαετίας του 50 και του 60 και ε, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της IPCC. Είναι η προβολή για την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα, επάνω αυτό το πράσινο. Κάτω βλέπουμε ε, τι έχει ε, αποφευχθεί από εκπομπές ε, χάρη στο πρωτόκολλο του Μαντρεάλ, ακριβώς γιατί δεν χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούμε λιγότερες ουσίες που εκπλέουν στη στιβάδα του Όσοντος. Και το 2010 οι επιστήμονες κατάφεραν να μετρήσουν και πραγματικά είναι στοιχεία τα οποία έχει χρησιμοποιήσει και ο καθηγητής Χάρης. Θα διαπιστώσετε ότι το 2010 καταφέραμε να μετρήσουμε τι αποφύγαμε. Οι σταθμισμένες εκπομπές και βλέπετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση, την πραγματική κατανάλωση το 2010 και την προβολή στο άλλο γαλάζιο τμήμα. Αυτή η διαφορά λοιπόν είναι πενταπλάσια με εξαπλάσια σε σχέση με το στόχο του πρωτοκόλλου του Κιώτο για την πλήρη συμμόρφωση μετά το 2020. Ναι, επισπεύδω. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Από το 1990 μέχρι το 2010 αυξήθηκε ο πληθυσμός της από 5 δισεκατομμύρια σε 7. Οι εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα ταυτόχρονα αυξήθηκαν από 20 σε 30 γιγατόνους. Η μείωση των ODS την ίδια περίοδο ήταν 10 γιγατόνι. Ε, σε σχέση με το 2010. Αυτές είναι οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Και 135 γίγατονς ε, εκτιμούν οι επιστήμονες ότι είναι η μείωση των ισοδυνάμων διοξιδίου του άνθρακα. Πολύ σύντομα να σας αναφέρω κάποια άλλα πολύ σημαντικά ευρήματα των ε, επιστημόνων που δρούν στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Μόνρεαλ και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι το όζον στη στρατόσφαιρα και η καταστροφή του και η κλιματική αλλαγή είναι ε, άρρηκτα συνδεδεμένες. Επίσης ε, και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η απορρόφηση ε, της υπεριόδους ακτινοβολίας. Όλα αυτά καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αποτελεί έβριμα των επιστημόνων μας. Αν συνεχίζαμε όπως το παρελθόν, η εκπομπή των υδοφρονανθράκων θα σήμαιναν 20% του συνόλου των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ε, 20%. 20% των συνολικών αποθεμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050. Ε, όχι το 20%, μέχρι 20%. Ναι, ναι, μέχρι 20%. Αλλά ξέρετε, είναι δύο τα στοιχεία. Το χαμηλότερο σενάριο είναι αυτό. Είναι 9 μάλλον και το υψηλότερο είναι 20. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, ναι, μέχρι 20%, όχι 20%. Εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τον αντίκτυπο στο κλίμα των ε, υδροφθορανθράκων, Διάφορα συμβαλόμενα μέρη πρότειναν μια τροποποίηση του πρωτοκόλου για να ελέγξουμε τους υδροφθοράθρακες. Διαβάζετε τις διαφάνειες. Τις διαβάζω και εγώ για να προχωρήσουμε γρήγορα. Λοιπόν, δύο είναι οι προτάσεις τις οποίες εξετάζουμε πάλι από αναπτυσσόμενες και απτυσμένες χώρες. Ε, για ε, να ελέγξουμε ε, τις HFC στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Επίσης για τη μείωση των και ζητούν παράλληλη εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιώτο και του Μοντρεάλ. Εξού και οι συνέργειες που λέγαμε σε επίπεδο εφαρμογής και σε επίπεδο πολιτικής. σε διάφορα επίπεδα γίνονται συζητήσεις, αλλά στο επίπεδο του πρωτοκόλου του Μόντρεαλ θα μπορούσαμε να βάλουμε οριακέ τιμές ε, που θα προστάτευαν σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα. Συμπέρασμα. Είναι βασικό παράδειγμα το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για μεσοπρόθεσμη και πραγματική δράση μετριασμού και συγκράτησης ε, της κλιματικής αλλαγής. Είδαμε ότι μέχρι 97% έχουμε μειώσει ε, παγκοσμίως τις ε, ουσίες που καταστρέφουν το όζο και επίσης καταφέραμε να μειώσουμε πάρα πολύ σημαντικά τους υδοφροράνθρακες. Για να προστατεύσουμε το κλίμα τα τελευταία 20 χρόνια. Και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι προτάσεις αυτές πραγματικά κινητοποιούν και τη βιομηχανία παγκοσμίω και ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε νέες εναλλακτικές τεχνολογίες. Τέλος, επιτρέψτε μου να τονίσω τα εξής δύο. Το πρωτόκολλο του Μόντρεγκαλ και το πρωτόκολλο του Κιώτο είναι ε, παγκόσμια σχήματα και καθεστώτα για την προστασία της ατμόσφαιρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις συνέργειες σε επίπεδο παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό. Το παγκόσμιο και το περιφερειακό σύστημα βοηθούν κανονικά, αποτελεσματικά και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ μπορεί να δώσει εμπειρία ετών, δύο δεκατιών για τη μείωση των διοξιδίων ε, και των αερίων και στην Ευρώπη έχετε μια πάρα πολύ ωραία σύμβαση, ε, τη γνωρίζετε, που έχει μειώσει και τα, τα οξύδια του θείου και τα οξύδια του αζότου και έχει μειώσει με επιτυχία την όξινη βροχή στην Ευρώπη. Επίσης, αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο θέμα και το μαύρο άνθρακα και τις πτυτικές ουσίες. Πώς τα λένε αυτά, τα πτυτικά συστατικά τα οργανικά, αυτό έψαχνα. Έτσι λοιπόν τα παραδείγματα αυτά επιτυχούς διεθνούς ε, ε συμφωνίας θα μπορούσαν να αντιγραφούν και να επεκταθούν και να συνεισφέρουν για μεγαλύτερη προστασία του κλίματος. Και αυτά τα καθεστώτα και αυτά τα σχήματα να συντονίζονται ακριβώς και να συνεργάζονται για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα παγκοσμίω και σήμερα και στο μέλλον. Ένα τελευταίο έχει να κάνει με την πρότασή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι κυβερνήσει και οι περιφέρειες δεν θα πρέπει να περιμένουν να συμφωνήσει η υδρόγειο ολόκληρη σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Υπάρχουν δυνατότητες σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν να προχωρούν μόνοι τους. η διακυβέρνηση, ε, ε, μάλλον οι κυβερνήσεις και οι περιφέρειες μπορούν να προχωρούν χωρίς να προχωρεί ταυτόχρονα η φίλιος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αυτό στέλνει το σωστό πολιτικό μήνυμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και άλλες χώρες συμμετέχουν και ρυθμίζουν μονομερός ή πολυμερός ή σε περιφερειακό επίπεδο τα θέματα αυτά. Και τα αέρια του θερμοκηπίου που επηρεάζουν, όπως είναι και ο μαύρος άνθρακας και άλλα που αναφέραμε προηγουμένως. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή, που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και πραγματικά στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα όχι μόνο στα κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά στον κόσμο όλο για το πόσο σημαντικό είναι να καταλήξουμε με ένα κοκτέιλ, ένα μείγμα πολιτικής ε, για μέσο πρόθεσμα ε, και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, well, thank you for that and thank you for... Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Όπως ξέρουμε με τα προβλήματα της εκπομπές από τις αερομεταφορές, ο ε, υπόλοιπος κόσμος συμφωνεί πάντα να κινείται πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι θα κινηθούμε σωστά σε αυτό το στάδιο. Ο Φίλιπ Οουέν είναι επικεφαλής μονάδας της Γενικής Διευθύνσεως για το Κλίμα, τη G-Clim. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει. Ευχαριστώ Λίντα, καλησπέρα όλοι, σε όλους σας. Όταν δει το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αισθανόμαστε κάποιε ανατριχίλε όταν μας τίθεται αυτό το ερώτημα. Χαίρομαι που ήρθα εδώ να σας πω τι κάνουμε, τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και να σα ικανοποιήσουμε, ελπίζω, με την απάντηση. Καταρχάς πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το πλαίσιο των στόχων μας. Τον Μάρτιο φέτος υιοθετήσαμε τον οδικό Χαρτί για το 2050 για μια οικονομία ανταγωνιστική με χαμηλή εκπομπή διοξίδιου του ανθρακό. Και στέσαμε φιλόδοξο στόχο 80% μείωση όσον αφορά τι οικιακέ εκπομπέ μέχρι το 2050, εν συγκρίση με το 1990. Και νέο οδικό χάρτη εστιάζεται βασικά στο διοξείδιο του άνθρακα. Εντό αυτού εμπεριέχονται δύο σαφεί τομεί που αναφέρονται σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Τι εκπομπέ άλλων αερίων, όχι διοξείδιο του ανθρακό. Πρώτα απ' όλα γεωργία Θέλουμε 42-49% μείωση στις εκπομπές μέχρι το 2050. Μη γεωργικός τομέας, μεθάνιο, φθοριού είχε αέρια, νητρικό, ε, αζωτούχα, οξύδια κλπ. Και θέλουμε μείωση 70-78% μέχρι το 2050. Εισαγάμε, θεσπίσαμε νομοθεσία πιο, για πιο βραχυπρόθεσμες περιόδους, καλύπτουμε εντός του ETS 3, 2013 με 2020, τα PFCs και τα οξύδια του αζότου ε, και έχουμε κάποιες βιομηχανικές εφαρμογές, ήδη έχουν αναφερθεί αυτές, ε, παρόμοια στην απόφαση για την κατανομή της προσπάθειας θέσαμε δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη-μέλη που κατά μέσο όρο μειώνεται έτσι η, ε, η, το διοξείδιο του άνθρακος μειώνεται, οξύδια του αζότου, μεθάνιο, SF6, PFCs, HFCs κατά 10% ε, το 2020 σε συγκρίση με το 2005. Για την περίοδο 2013 με 2020 μιλάμε. Η απόφαση για την καταναμή της προσπάθειας ε, εξετάζει την καύση καυσίμων, ε, απομάκρυνση από τα παραδοσιακά καύσιμα, ε, τι γίνεται με τα απόβλητα, με τη γεωργία, την χρήση διαφόρων διαλυτικών ουσιών κλπ. Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και απηχούν τα στοιχεία αυτά που ανέφερε μόλις τώρα ο Μάρκο όσον αφορά το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που υπήρξε επιτυχέστατο και συμφωνώ ότι ήταν επιτυχέστατη η Διεθνή Συμφωνία και υφίσταται από το τέλος δεκαετίας του 80 και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Είδαμε σημαντική μείωση των ουσιών που μειώσει τη βάδα του όζοντος, 97% μείωση των ουσιών αυτών. Αυτό αντιστοιχεί σε 135 γιγατών διοξιδίου του άνθρακος μεταξύ 1990 και 2010 και αυτό είναι για όλο τον κόσμο το στοιχείο. Υπήρξε όμως που θεσπίστηκε ευρωπαϊκή νομοθεσία από την δεκαετία του 90 και συμμετείχε στην προσπάθεια η Ευρώπη. Αυτό είναι σαφέ. Παρομοίω, έχουμε μειώσει τι εκπομπέ του μεθανίου από άμεσε εκπομπέ στον τομέα των αποβλήτων κατα... μειωθήκαν κατά 10% από το 1995 μέχρι το 2007 και για τις χωματοερές είδαμε έχουμε μείωση 20 μεγατόνων το χρόνο σε αντιστοιχεία διοξιδίου του άνθρακος τα πρόσφατα χρόνια, τελευταία χρόνια. Έχουμε και τον κανονισμό για τα θεωριούχα αέρια. Ε, εφαρμόστηκε το 2006 η νομοθεσία. Πλήρως το 2008 και σε όλους τους τομείς το 2010. Και είδαμε μειώσεις όσον αφορά τον κανονισμό για τα διάφορα αέρια και την οδηγία για, τους, ε, για τα κινητά κλιματιστικά. Πρόσφατα τέθησε ισχύ, αλλά ελπίζουμε ότι τελικά μπορούμε να περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες ε, μειώσεις στου αφορά τις εκπομπές. Ένας τομέας είναι η αναθεώρηση του κανονισμού για τα αυθοριούχα αέρια. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τι γίνεται το 2011. Θα εκτεθεί μια έκθεση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φθινόπωρο. Θα αναφέρεται στην εφαρμογή, πώς χειρίστηκαμε την εφαρμογή της νομοθεσίας, ποιο είναι το διεθνές πλαίσιο και ποιες περαιτέρω επιλογές μπορεί να υπάρξουν και περαιτέρω μελέτη, ε, κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε αν θέλουμε να υποβάλουμε νομοθετικού περιεχομένου πρόταση το 2012. Μία επιλογή σαφώς είναι να μην κάνουμε τίποτα, όμως αυτό δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο δοθέντων των στόχων που προαναφέραμε όσον αφορά τον οδικό χάρτη για το διοξείδιο του άνθρακος. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην ε, ε, πιστοποίηση, ορόφηση, κατακράτηση να διατηρήσουμε κάπως το status quo θα μπορούσαμε να πετύχουμε, αλλά ίσω θα θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι δεν αρκούν αυτά τα μέτρα, ίσως θα πρέπει να δούμε μια εναλλακτική λύση. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσει. θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αξιολόγηση του αντικτύπου, αλλά υπάρχει ένα τομέα που θα πρέπει να αντιληφθεί περαιτέρω, αλλά και στο παγκόσμιο πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα HFC στο πρωτόκολλο του Μοντρεάλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ενεργή όσον αφορά την υποστήριξη ε, της προτάσεις της Μικρονησίας και της Βορείου Αμερικής και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 28 συνολικά κράτη της Ευρώπης, υπέγραψαν τη δήλωση, τη διακήρυξη που διατυπώθηκε στο τέλος της συνόδου της Μπανκόκ το περασμένο φθινόπωρο. Παράλληλα λοιπόν με τα θωριούχα αέρια εξετάζουμε και το μεθάνιο υπάρχει νομοθεσία για την ανακύκλωση 50% των δημοτικών αποβλήτων και 50% των οικοδομικών αποβλήτων μέχρι το 2020. Έτσι θα μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές στον τομέα αυτό, να μειωθούν, να μειωθεί και, η, και τα απόβλητα τα βιοδιασπόμενα σε αυτή την περίοδο. Οι εκπομπές από τη Γεωργία μειωθήκαν κατά 20% από το 1990 μέχρι το 2006 και είναι ένα κλειδί για την πρόοδο. Εκπομπές του μεθανίου είναι μεγάλο ποσοστό ε, εκπομπών της Γεωργίας και προσβλέπουμε στον οδικό χάρτη αυτών για τη μείωση ε, αυτών των εκπομπών μέσω πολλαπλής συμμόρφωσης, ε, γεωργική χρηματοδότηση κλπ. στα πλαίσια δημοσιονομικών προπτικών από το 2013 και πέρα και θέλουμε να ακολουθήσουμε και άλλες ιδέες πιο αποτελεσματική χρήση των διαφόρων υπασμάτων, ταξινόμηση των βιοκαυσίμων, άλλες μορφές πιο βιώσιμης γεωργίας και νομίζω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για την βιοοικονομία από τη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία τον επόμενο χρόνο. Βλέποντας τώρα τι γίνεται με την τροπόσφαιρα, το άνθρακα ε, και το όζον. Ε, από το 2008 έχουμε την οδηγία για την ποιότητα σφαιρικού αερίου και μειώνει τα PM10 και PM2,5. Έχουμε οριακές τιμές και στόχους ήδη. Ε, είναι δύσκολο να πετύχουν στόχους στα κράτη-μέλη και σίγουρα έχουν δοθεί παρατάσεις σε κάποιες περιόδους όσον αφορά το όριο του 2010 για την ε, συμμόρφωση. Πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει τη θεματική στρατηγική για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και θα εξετάσουμε πλέον το θέμα του μαύρου άνθρακα και το όζον σε επίπεδο εδάφους και άλλους ρηπαντές της ατμοσφαίρας. Αναφέρθηκε ο Μάρκος στη σύμβαση για τη συνοριακή ρήπανση της ατμόσφαιρας Είμαστε πολύ δραστηριοποιημένοι στον τομέα. Εξετάζουμε και το μαυράνθρακα και το τροποσφαιρικό όζον. Εν κατακλείδη, λοιπόν, έχουμε τον δικό χάρτη για το 2050 με σαφείς στόχους. Έχουμε νομοθεσία που ήδη φίσταται για να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων του 2020. Έχουμε διάφορα θέματα πολιτικής με τα φθοριούχα αέρια και με την ε, ποιότητα του σωρικού αέρα Παραμένει όμως μια πρόκληση πρέπει να καλυφθεί. Αυτή η πολύ ψηλοί ε, στόχοι που έχουν τεθεί για το 2050 πρέπει να εξεταστούν εκ του σύνεγγυ στα επόμενα χρόνια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι θα πετύχουμε αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Okay, we... Καλώς. Ακούσαμε τρεις εξαιρετικούς ομιλητές και τώρα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Όχι μόνο βουλευτές και άλλοι συνάδελφοι. Ο Βιτόριο Πρόντι βλέπω πρώτος στην ερωτήση. Um, black carbon, uh, Για το μαύρο άνθρακα. Σωστά είπατε ότι η περίοδος ζωής στην τροπόσφαιρα είναι λίγες μέρες, ε, λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως σημαντική συγκέντρωση, ε, εικάζεται, στη στρατόσφαιρα. Αλλά δεν υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί ε, για να καταλάβουμε πώς ε, παράγονται οι βροχοπτώσεις εκεί. Είναι ανοιχτό ακόμα το πρόβλημα και συνδέεται άμεσα με την άμεση υπερθέρμανση της στρατόσφαιρας. Διότι στη στρατόσφαιρα, εξ όσων θυμούμε, παραμένουν τα αέρια χρόνια ολόκληρα. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και πάντα προβληματίζομαι και αναρωτιέμαι. Δεν θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, να κάνουμε ένα πείραμα. Τι γίνεται σε περίπτωση καταστροφικής υπερθέρμανσης. Ε, ε, κάπως να προσωμιώσουμε ας πούμε ηφαιστειακές εκρήξεις. Διότι νομίζω ότι ε, θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Να αυξήσουμε τη θερμοκρασία, ας πούμε, με άμεση ε, έγχυση σωματιδίων στην στρατόσφαιρα. Για να έχουμε κάποια ιδέα τι θα γίνει αν υπάρξει τόσο καταστροφική υπερθέρμαση; Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτά τα ε, ακραία φαινόμενα. Στο τέλος θα να μας πείτε ποια είστε και ε, ποιον εκπροσωπείτε. Νατάσα Χέλη από την Υπηρεσία Ερευνών ε, Περιβάλλοντος συμμετέχω και ε, τις τελευταίες δεκαετίες στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε διάφορες ε, συσκέψεις ενεχομένων ε, για τα αέρια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Όουεν, στις διαφάνειες μας δείξατε διάφορες ε, Εναλλακτικέ λύσεις για βελτίωση της νομοθεσία, Μείωση των υδροφλωρανθράκων είπατε για τα αέρια που περιέχουν θόριο. Και μετά αναφερθήκατε και στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Υπάρχει συνένεση για τη σημερινή νομοθεσία, για το σημερινό κανονισμό και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται. Αν λέτε διεθνώς ότι σταδιακά θα πρέπει να εγκαταληφθεί είναι μικρότερη φιλοδεξία ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς αντισταθμίζεται. Ο Συμπρόεδρος έχει ερώτηση. Μια απλή ερώτηση θα είχα εγώ, λέει ο κύριος Κυλακάκης, και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι στη φυσική ε, αναζητούμε την ενιαία ε, θεωρία, η θεωρία των κβάντων ας πούμε, πώς ε, συγκεράζεται με τη κλασική φυσική. Εσείς σκέφτεστε καμιά ενοποιημένη θεωρία έτσι ώστε εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και μη διοξιδίου να συνενωθούν για να γνωρίζουμε εμείς που κάνουμε πολιτική πόσο θα κοστίσει αν θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μας, τι μέσα. Μπορούμε να έχουμε μια συνολική σφαιρική προσέγγιση ε, των αερίων το διοξίδιο και αυτό που δεν είναι διοξίδιο. Γιατί έχω δει πολλές διαφορετικές πολιτικές και μέσα πολιτικής, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος για μας να κρίνουμε αν κάνουμε καλή δουλειά ή όχι. And I have a question for this round. just, um, Και εγώ έχω ερώτηση. Μιλήσαμε για περικοπή των HFCs και τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων είναι μεγάλη πηγή αυτών των θεωρών θράκων ε, και σωματιδίων. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο στον τομέα. Διότι πιθανότατα θα πιέσει η βιομηχανία να μην κάνουμε περισσότερα. Ποιο μπορεί να επηρεαστεί από τα μέτρα, αν κάνουμε περισσότερα. Ποιο θα είναι τα, ποια θα είναι τα λόμπι που θα μας προσεγγίσουν πρακτικά. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά. Φίλιπ, είχε μια διαρωτήση που απευθύνθηκα σε σένα. Και ο δόκτωρ χάρη ίσω να είναι και όσο πρέπει να απαντήσει στον ε, κύριο Πρόντι. Ο Φίλιπ πρώτο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρο ε, σε ποιον απευθύνω την τελευταία ερώτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ξεκίνη. Έτσι. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω τουλάχιστον. Ε, Καλώ. Με αντίστροφη σειρά. Όσον αφορά τι εκπομπέ. Ο μαύρο άνθρακα, από ό,τι γνωρίζω, ξέρω λίγα, προέρχεται από πολλέ πηγέ. Από τα οχήματα και βιομηχανικέ ε, εφαρμογέ εν γέννη. Θα πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται με την νομοθεσία την ποιότητα της ατμόσφαιρας, εθνικές οροφές όσον αφορά στις εκπομπές, ε, οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας κλπ. Υπάρχει ήδη νομοθεσία που προσπαθεί να μειώσει αυτές τις εκπομπές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τα οχήματα. Είναι μια πρόκληση όσον αφορά ε, την εκ των υστέρων εγκατάσταση διάφορων ανταλλακτικών και εξοπλισμό. Και δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση στο να μπει κάποιο εξοπλισμό σε παλιό όχημα. Είναι δύσκολο ερώτημα αυτό. Ε, άλλο θέμα. Ότι όλα αυτά πάνε στην ατμόσφαιρα. Και γι' αυτό ενδιαφέρονται οι συνάδελφοί μου του περιβάλλοντος, ενδιαφέρονται για τη σύμβαση για μακροπρόθεσμη διασυνοριακή ρήπανση της ατμόσφαιρας. Και θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό το τομέα για να περιορίσουμε την ε, θάλη των μαυρών άνθρακα, δηλαδή στο μέτρο του δυνατού. το ερώτημα της ε, υπηρεσίας περιβάλλοντος, ε, προστασίας περιβάλλοντος δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση. Ήμασταν πολύ δραστηριοί για να υποστηρίξουμε την μείωση των HFCs πέρσι, σύμφωνα τάσεις των βορειοαμερικανικών χωρών και της Μικρονησίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει και τις δύο πρωτοβουλίες και φέτος και στο Μοντρεάλ τον Αύγουστο και στον Παλί ε, τον Νοέμβριο στις δύο συνεδριάσεις του πρωτοκόλου του Μοντρεάλ. Και είμαστε αρκετά ενεργοί, είμαστε στο ένα τρίτο των χωρών που έχουν ήδη υπογράψει αυτή την, ε, αυτό το πρωτόκολλο. Και χρειαζόμαστε και χρόνο βέβαια για να εξετάσουμε τις διάφορες δυνατότητες που έχουμε στην Ευρώπη. Να κάνουμε τίποτα ή να βελτιώσουμε τα μέτρα συγκράτησης να δούμε τι γίνεται με απαγόρευση, σταδιακή εξάλληψη διαφόρων ε, ε, μεθόδων που παράγουν ε, τα αέρια. Είναι δουλειά που θα συνεχιστεί. Η έκθεση για την εφαρμογή της νομοθεσίας θα υποβληθεί τον, το φθινόπωρο και εν ευθέτω χρόνο μετά από ίσως εξ, ικανοποιητική αξιολόγηση συνεπιών θα έρθουμε μετά στο θέμα του κόστους που έθεσε ο κύριος Σκυλακάκης. Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν το 2012 κάπως. Τώρα, το να εξετάσουμε μαζί, ολιστικά αυτά τα αέρια, είναι ενδιαφέρον. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι ήθελα να κάνω, έκανα κάποια έρευνα η σημερινή παρουσίαση και με ενδιαφέρε πολύ να καταλάβω τι γίνεται, ε, πώς μπορεί να συνεργαστούν όλες αυτές οι διαφορετικές πολιτικές. Και με ικανοποίησε αυτό που είδα. Εστιαζόμαστε βασικά στο πλαίσιο Κιώτο για τα αέρια και στο ETS και για τις αποφάσεις που λάβαμε εκτός ETS. Αν θέλετε τα στοιχεία, τα στοιχεία θα είναι αξιολόγηση αντιχτύπων για τις νομοθετικές πράξεις. Άρα εκεί συμπεριλαμβάνεται και το κόστος. Υπάρχουν, θα υπάρχουν οι πληροφορίες που θέλετε. Είναι πολύ χρήσιμο να γίνει και αυτή η σύνοδος που συνοψίζουμε, να δούμε τι γίνεται στη Γεωργία, τι γίνεται όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, να δούμε τη γενικότερη εικόνα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ο καθηγητής Χάρης έχει τον λόγο. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το μαύρο άνθρακα ε, που πάει στη στρατόσφαιρα. Καλό είναι που πάει στη στρατόσφαιρα για τους εξής δύο λόγους. Μάλλον έχει δύο δρόμους, από τους τροπικούς, από τη μια και από την άλλη. Όταν έχουμε μεγάλες δάσοπυρκαγιές, υψώνονται πάρα πολύ ψηλά μέχρι τη στρατόσφαιρα τα ε, σύννεφα καπνού. Οι αερομεταφορές δεν ε, εκπέμπουν τόσο πολύ ε, εθάλη, ε, ίσως στους τροπικούς που είναι πιο εύκολο να ανέβει στη στρατόσφαιρα. Προσωπικά θα έλεγα ότι ε, αυτό το καιρό γίνεται έρευνα για τον αντίκτυπο, διότι το όζον και τα αεροσόλα από θιούχα ε, ε, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, αυτά είναι που κυριαρχούν και όχι τόσο οι εθάλοι και τα σωματίδια στη στρατόσφαιρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο έχουμε συμπεράσματα της έρευνας. Ε, είναι ενδιαφέρον να το ψάξουμε ακριβώς ερευνητικά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Το πείραμα για την καταστροφή, δηλαδή να στείλουμε μαζικά σωματίδια εθάλης, γεωμηχανικής ας πούμε, ξέρω ότι γίνονται τέτοια πειράματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού με άμεση έγχυση τέτοιων σωματιδίων στη στρατόσφαιρα με τρόπους πάρα πολύ ευρηματικού αυτή τη στιγμή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζω το πείραμα που γίνεται. Κυρίως οι μηχανικοί ψάχνουν πώς θα στείλουν στη στρατόσφαιρα τόσα πολλά σωματίδια. Ξέρετε ότι είναι 18 χιλιόμετρα ε, στους τροπικούς για να το κάνουμε. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογία ε, για να δούμε ποια θα είναι η ατμοσφαιρική επίπτωση, ας πούμε, ο αντίκτυπος. Υπάρχουν θέματα πολιτικά και δεοντολογικά και κοινωνικά. Και αυτή τη στιγμή αποκτήσουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, θα δούμε. Σε ό,τι αφορά τη γεωμηχανική, είναι ε, και αυτό ένα ζήτημα για να στείλουμε σωματίδια στη στρατόσφαιρα. Είναι πολύ επίμαχο. Πάντως οι πάντες συμφωνούν ότι πριν το κάνουμε θα πρέπει να το μελετήσουμε πάρα πολύ καλά, να το ψάξουμε ερευνητικά, να, το έχουμε ας πούμε στην κολότσεπη αν θέλετε ως εναλλακτική λύση, αλλά δεν θα το αναλάμβανα ως πείραμα αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να προσθέσω μερικά πράγματα για την Εθάλη και το μαύρο άνθρακα και τις επιπτώσεις, όχι στην Ευρώπη, ε, αλλού η μεγάλη πηγή είναι ε, το μαγείρεμα με, με ξύλα, με, κάρβουνα στην Ήπεθρο, στην Ανατολική Ασία, νομίζω και στην Νότια Αμερική. Και είναι ξύλο, έχουν αλλάξει τις ε, πρακτικές τεχνολογικά, αλλά στην νότιο Ανατολική Ασία το μόνο που σταματάει ε, μάλλον το, ε, είναι τα Ιμαλάια. Αν, αν το σταματήσουμε να βγαίνει στη στρατόσφαιρα θα σταματήσει να πηγαίνει και στα Ιμαλάια και να λιώνουν οι πάγοι και να αλλάζει το κλίμα. Σας είπα τι επίπτωση έχει αυτό κοντά σε λευκές επιφάνειες, σε παγετώνες και σε μέρη που καλύπτονται από χιόνι και από πάγο, ας πούμε τα Ιμαλάια. Κάτι άλλο και ένα προσωπικό σχόλιο τώρα γενικότερα από κάποιον που δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων πολιτικής. Αν κάποιος λαμβάνει μονομερή δράση, για μένα θα ήταν ε, σωστό και ειλικρινές να είναι διακλαδική η ε, αντιμετώπιση. Και είναι σωστό αυτό, αλλά όταν αρχίζει κανείς να αποφασίζει πολυμερός, χρειάζεται κάποια ισορροπία γιατί ε, κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικά συμφέροντα από εσά και έχουν διαφορετικές σκέψεις για το κόστος και την ωφέλεια. Ενώ εσείς όταν παίρνετε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά την Ευρώπη αυτό. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο Μάρκο ότι πραγματικά ε, πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις και τοπικές και περιφερειακές και παγκόσμιες. Να μην περιμένουμε μόνο τις παγκόσμιες. Αυτό που είπε ο Μάρκο για τους Ε, είδαμε να μειώνονται και στη Βόρεια Αμερική και στη Σκανδιναβία. Και οι εκτιμήσεις για ε, το ότι ε, κερδίζουμε είναι δύο ή τρεις φορές περισσότερο από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Γιατί, Γιατί αυτοί άρχισαν από το 1970 και μετά να αναλαμβάνουν τέτοιε δράσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι η δράση τοπική, περιφερειακή και αργότερα παγκόσμια. Έχετε τίποτα να προσθέσετε, να τα προσθέσετε. Καλώς. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε ερωτήσεις. Ο κ. Κυλακάκης λοιπόν θα κλείσει αυτό το στάδιο της συζήτησης. Νομίζω ότι τώρα γνωρίζουμε καλύτερα την περιπλοκότητα του θέματος, διότι έχουμε πολλά διαφορετικά αέρια, πολλές επιρροές, πολλά μέσα πολιτικής και χρειαζόμαστε πολύ ακόμα δουλειά στο Κοινοβούλιο σαν νομοθέτες για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε πολιτικές που μας ικανοποιούν θα συμφωνούσα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει αν κινείται μονομερός. Στη δική μας περίπτωση, μονομερής κίνησης δεν θα είναι επιτυχή στο τέλος. Χρειαζόμαστε πολυμερή προσέγγιση. Όσο πιο περίπλοκη είναι η διαπραγμάτευση, τόσο πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν όλοι περί τίνος πρόκειται και όχι μόνο αυτό, αλλά και ποιε είναι οι πραγματικές επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάμαι εδώ και μερικά χρόνια, πέντε χρόνια νομίζω, ο Νίκολας Σταν ε, έδωσε την αναθεώρησή του. Είχε τεράστιο αντίκτυπο όσον αφορά το πώς βλέπαμε την αλλαγή του κλίματος άλλαξε η άποψή μας μετά την αναθεώρηση αυτή. Μας άλλαξε. Γιατί ενοποιούσε τα διάφορα στοιχεία. Ήρθε η ώρα νομίζω να ξανανοίξει αυτή η αναθεώρηση μετά από πέντε χρόνια. Αυτή η έκθεση, αυτή η ανάλυση. Να προσθέσουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ανάλυση, γνώση σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακος και όχι μόνο, και όσον αφορά και τις άλλες ουσίες, όσον αφορά την καινοτομία και το τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε πολλά περισσότερα και όλα αυτά τις γνώσεις που έτσι μαζέψουμε. Και στο Κοινοβούλιο αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε και ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες τη βοήθειά τους, κυρίως τους εκπροσώπους του πρωτοκόλου του Μοντρεάλ. Τους βλέπω σαν φάρο επιτυχίας. Και αυτό σπανίζει σε πολυμερείς προσπάθειες. Πρέπει να πάτε στη Βόρεια Αμερική να τους μιλήσετε για την πολυμερή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, once more heartily welcome. We are coming now to the second part of our seminar organized by our policy department on this non-CO2 climate. Και ερχόμαστε στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου μας. Έχουμε εδώ την κυρία Σάτου Χάσο από τους Πρασίνους. Πολύ σημαντικό αυτό που αναλάβαμε διακομματική πρωτοβουλία από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και πραγματικά θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα για να συμφωνήσουμε. Panel, uh, there are Uh, όπως είδαμε και στην πρώτη ενότητα, τα αέρια του θερμοκηπίου επηρεάζουν πάρα πολύ το κλίμα μας. Ε, θα πρέπει να είναι σφαιρική ενιαία η ε, αντιμετώπιση, όπως είπε και ο κύριος Κυλακάκη. Αλλά έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και τώρα στο δεύτερο πάνελ έχουμε εκπροσώπους ακριβώς ε, που θα μας μιλήσουν για αυτή τη διάσταση, τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Παρακαλώ παρακολουθείτε την ελληνική διερμηνία. Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε τα ελληνικά, αρκεί να μας κάνετε ένα μικρό νόημα. Είμαστε πίσω από το Προεδρείο, να ακούτε ελληνικά σας παρακαλώ πολύ.